Οπότε, έκθεση Άρα, Αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, θα κάνουμε πολλά πράγματα για πρώτη φορά. Σήμερα το πρωί έλαβα πολλά τηλεφωνήματα. Σας είδα, σας είδα. Για αυτή την ψηφοφορία σας είδα. Σας διαβεβαιώ ότι ήρθα με το αυτοκίνητο ε, θα φύγω αύριο. Έχω όλο το χρόνο στη διάθεσή μου. Επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο μέσω του κανονισμού να γίνουν ψηφοφορίες ε, με μπλοκ ψηφοφοριών. Αλλά φυσικά οι υπηρεσίες θα καθορίσουν, θα προετοιμάσουν αυτές τις, ε, αυτά τα μπλοκ. Ξέρω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για αυτά, οπότε θα πρότεινα στην αρχή να αρχίσουμε την ψηφοφορία και μετά από λίγο χρόνο θα σας ρωτήσω εάν πραγματικά θέλετε να ψηφίσετε κάθε μεμονωμένη τροπολογία ή, θα ή αν θα μπορούσαμε να κάνουμε ψηφοφορία σε μπλοκ. Διαδικαστικό εσείς παρακαλώ κύριε. Η κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το θέμα δεν είναι ο χρόνος. Το θέμα είναι να έχουμε ένα καλό νομοθέτημα μετά την ψηφοφορία. Αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ότι έχουν οπαδοποιηθεί οι τροπολογίες με τα ονόματα των συντακτών των τροπολογιών. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το νομοθέτημα που θα προκύψει δεν θα είναι καλό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις θέσεις εργασίας και εμείς θα γίνουμε περίγελος. Έτσι λοιπόν ζητάμε μια έναν κατάλογο ψηφοφοριών που να έχει προετοιμαστεί σωστά. Έχουμε 1.400 τροπολογίες, θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε έναν κατάλογο ψηφοφοριών για το Στρασβούργο. Έτσι λοιπόν απευθύνω έκκληση σε όλους να υποστηρίξετε το αίτημα αυτό. Λοτόφσκι. Πρόεδρε, από πλευράς ομάδας ECR προτείνω να αναβληθεί η ψηφοφορία αυτή γιατί η αλληλουχία των τροπολογιών παραβιάζει το 194.2 και 8 του εσωτερικού μας κανονισμού. Υπάρχουν δύο εναλλακτικέ λύσεις. Έχουμε ταυτόσιμες τροπολογίες που είναι σε διαφορετικά μπλοκ και θα, αν το ψηφίσουμε έτσι δεν τηρούμε το 194-9 του ιστορικού κανονισμού. Έχουμε βρει τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις, γιατί αυτά τα μπλοκ τροπολογιών έχουν συσταθεί με βάση τους συντάκτες των τροπολογιών και όχι με βάση το περιεχόμενο των τροπολογιών. Και αυτό είναι απόλυτα αντίθετο με μια σωστή διαδικασία. Οπότε, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μέσα αυτής της διαδικασίας να κάνουμε σοβαρό διαδικαστικό λάθος και μπορεί γι' αυτό να γίνουν προσφυγές στα δικαστήρια. Για τρίτη φορά κατά δεν τρέχουσα θητεία. Οπότε κάνω έκκληση να στηρίξετε το αίτημά μου για αναβολή. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Πολύ ευχαριστώ. Εάν όμως είχατε την καλοσύνη, αντί να διαβάζετε έτοιμες από πριν ομιλίες, να ακούγατε τι έχω πει, δηλαδή ότι πρόκειται να ψηφιστεί αυτό το αίτημα. Η κυρία πριν από εσά έκανε το ίδιο αίτημα για αναβολή και ως εκ τούτου, χωρίς να θέλω να ε, επιμείνω περισσότερο, θα προτείνω να ψηφίσουμε τώρα. Ψηφίσαμε και χτες, άλλη μια φορά τώρα λοιπόν, υπέρ της αναβολής παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Εξακόσια παρακαλώ υπέρ κατά Αποχές απερίφθη 630. Όχι, ζητώ συγγνώμη. ...645, 691, 650 και λοιπές τροπολογίες που προτείνουν την απόρριψη ονομαστικά. Παρακαλώ. Ψηφίσατε. Πέρασε. Και έτσι πάω στην 629 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 630. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε πολύ καλά ότι μετά γίνεται το αίτημα για την επαλήθευση θα κάνω ό,τι μπορώ σήμερα για να επιφυλάξω ομαλέ κοινοβουλευτικέ διαδικασίε, αλλά δεν θα επιτρέψω και σε κανένα να παρεμποδίσει τι ψηφοφορίε. Και παρακαλώ να μην υπερβάλλετε. Deshalb lasse ich das jetzt zunächst mal überprüfen. Άρα κάνουμε έναν έλεγχο. Άρχεται παρακαλώ η ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται και χρειάζεται πλειοψηφία των 2 ε, τρίτων. Να το έχετε αυτό υπόψη. Βέβαια είναι ξεκάθαρο, ε, το αποτέλεσμα δεν θα ζητώ πάλι. 6.30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εντάξει, ελέγχουμε την 630, άρχεται η ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 631 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 632. Να ελέγξουμε την 631. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφεται και εδώ με την πλειοψηφία των δύο τρίτων. Θέλετε το λόγο της διαδικασίας. Ναι. Για διαδικαστικό ήθελα το λόγο. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο και θα πρότεινα να συνεχίσουμε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, δυνατόν. Μου επιτρέπετε κυρία Γκραπίνη να το αποφασίζω εγώ αυτό. 633 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 633 λέω τώρα πρόεδρος. 634 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 635 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 618 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 619 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 620 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 621 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 622 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 623 ψήφι υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 624 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 625 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 626 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 627 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 628 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 636 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 637 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 638 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 631 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 640 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 641 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 642 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 643 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 644 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ολοκληρώσαμε την πρώτη δέσμη, αγαπητοί συνάδελφοι. 1100 συνολικά τοπολογίες. Περνάμε στην δέσμη Β και προχωρούμε 763 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 292 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 293 ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 294 ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 295 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 296 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Le ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 297 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι όλοι πέρα Απορρίπτεται. 2.98 ψήφι περ. Κατά. αποχε Απορρίπτεται. 2.99 ψήφι περ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 300 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα. Απορρίπτεται. 301 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 302 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 303 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 304 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 222 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 224 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 225 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές από 226 ψήφοι κατά αποχές απορρίπτεται 227 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 228 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 229 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 230 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 232 ψήφι υπέρ κατά αποχές 2, 72-33 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απο 2, 72-34 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.35 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 2.36 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 2.38 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 2.39 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 2.40 ψήφι υπέρ, κατά αποχές το 241 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 242 ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται 243 ψήφι υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 2.44 ψήφι υπέρ, κατά αποχές το 2.45 ψήφι υπέρ, κατά αποχές το 2.46 ψήφι υπέρ, κατά αποχές το 2.47 ψήφι υπέρ, κατά αποχές από 48, ψήφι υπέρ κατά αποχές από 49, ψήφι υπέρ κατά αποχές από 50, ψήφι υπέρ κατά αποχές από 251, ψήφι υπέρ κατά αποχές από 252, ψήφι υπέρ κατά αποχές από 253, ψήφι υπέρ κατά αποχές από 254, ψήφι υπέρ κατά αποχές από 255, ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 256 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 257 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 258 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 259 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 260 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Αγαπητοί συνάδελφοι, Δεν μπορώ να πάω πιο γρήγορα, δεν μπορείτε ούτε εσείς πιο γρήγορα, ούτε και οι διερμηνείς μπορούν πιο γρήγορα. Και επειδή έτσι όπως παρατηρώ τελευταία ε, υπάρχουν πολλές, πολύ μεγάλη διαφορά από 550 έως 2 τρίτα ψηφίστε υπέρ συνήθως, οπότε το σκέφτομαι μήπως τελικά ε, να ακολουθήσω την ε, υπόδειξή σας να ψηφίσουμε ομού. lassen sie uns zwei drei minuten zeit in diese frage ε, δώσουμε δύο-τρία λεφτά στο να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Κύριε Μαρινέσκου. Dear colleague, dear Vice President. Κύριε Διπρόεδρε, άκουσα το αίτημα των συναδέλφων από την αρχή, αλλά αυτό που ψηφίζουμε δεν αφορά το περιεχόμενο. Αφορά περιφερεια... τα... την αντιπαράθεση της περιφέρειας σε σχέση με, την... με τον πυρήνα. Άρα, ας ψηφίσουμε άρθρο προς άρθρο, παράγραφο προς παράγραφο, στο περιεχόμενο δηλαδή. Γιατί δεν πρέπει να ψηφίζει έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να ψηφίζουμε ανα ομάδες ε, τροπολογιών είναι ότι υπάρχουν ομάδες ε, βουλευτών που πρότειναν τροπολογίες. Σε ένα μπλοκ υπάρχει, ας πούμε, τροπολογία για το άρθρο 4, 9, 12, που είναι άσχετες μεταξύ τους. Απ' τη μία μιλάμε για την, το χρόνο οδήγησης, για την ηλικία του οδηγού, για το που παρκάρει το φορτηγό του κτλ. Καμία σχέση. Άσχετες τροπολογίες δηλαδή θα, θα ψηφίσουμε μαζί. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν ακολουθούμε τους κανόνες του Κοινοβουλίου. Φταίνε οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου για αυτό το χαμό που δημιουργήθηκε. Κύριε Μαρινέσκου, όλα αυτά που είπατε τα ακούω, αλλά ε, αποκρούω αποφασιστικά την τελευταία σας πρόταση. Ε, κύριος Λαμπέρτς, ε, Πρόεδρε, ακούω αυτό που λέει ο κύριος Μαρινέσκου, ότι ομαδοποιήσαμε ε, βάσει των συντακτών της ε, Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά ακριβώς οι ομάδες ε, των τροπολογιών έχουν μια πολιτική λογική. Δηλαδή, οι διάφορες ομάδες των συντακτών των τροπολογιών το έκαναν έχοντας μια καθολική εικόνα το άρθρο, ε, και, μάλλον την, ε, της έκθεσης βέβαια σε διάφορα άρθρα, αλλά έχουν πολιτική συνάφεια και συνοχή μεταξύ τους συντροπολογίες, οπότε έχει νόημα να τις ψηφίσουμε ομαδών. Ωραία. Ακούσαμε τις δύο απόψεις προσωπικά. Θεωρώ, κύριε Μαρινέσκου, ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να γελιοποιείται και από διάφορες κατευθύνσεις. Μπορούμε να γελιοποιηθούμε και ψηφίζοντας σαν μπλοκ, αλλά και ε, ακολουθώντας τη διαδικασία που ε, ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Το θέμα είναι να βρούμε μια αντικειμενική λύση που να εξυπηρετεί το σκοπό μας. Έχουν γίνει κάποιες προεργασίες ε, στην Επιτροπή, την αρμόδια, που πρέπει να ληφθούν και αυτές υπόψη. Και τίνω να συμφωνήσω περισσότερο με τον συνάδελφο Λάμπερτς. Και σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού έχουμε τη δυνατότητα να ομαδοποιούμε τις τροπολογίες και υπάρχει και αποχρό λόγος γι' αυτό. Και θα δώσω λόγο στον κύριο Κόρμπετ που φέρει και την κύρια ευθύνη του κανονισμού. Ομολογώ, Πρόεδρε, ότι εγώ συνέταξα αυτή την παραγραφό του εσωτερικό κανονισμό και υπάρχει εδώ και χρόνια αυτή η διάταξη. Υπάρχει ακριβώς για να προβλέψει τέτοιες καταστάσεις, όπου έχουμε ασυνήθιστο αριθμό τροπολογιών και μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις τροπολογίες όπως ακριβώς περιέγραψε ο κύριος Λάμπερτς ή με άλλους τρόπους, με λογικό πάντα τρόπο, ούτω ώστε να μπορέσει να εργαστεί σωστά το Κοινοβούλιο με σεβασμό των απόψεων των βουλευτών. Έχει νόημα να ομαδοποιήσουμε τις τροπολογίες με αυτόν τον τρόπο και θα μας επιτρέψει να εργαστούμε αποτελεσματικά χωρίς να χάσει κανένας βουλευτής το δικαίωμά του να υποβάλει τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Κόρμπετ. Λοιπόν, δεν θα δώσω το λόγο τώρα για διαδικαστικό και επί του κανονισμού σε κανέναν. Ακούσαμε δύο απόψεις και μία εξήγηση. Θα μπορούσα να το αποφασίσω μόνος μου. Και ε, άφησα να νεωθεί ότι συμφωνώ με τον κύριο Λαμπέρτς. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω εσάς, συμφωνείτε να ψηφίσουμε ομαδικά τώρα τις τροπολογίες. Μπλοκ, ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Das lasse ich überprüfen. Die... Ας το ελέγξουμε παρακαλώ, άρχεται ηλεκτρονική επαλήθευση. alle Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Με πλειοψηφία δύο τρίτων, αν είναι σωστή υπολογιστή μου. Άρα, ε, το μπλοκ Β, λοιπόν, συνεχίζουμε από την 261 μέχρι ε, την 332. Ε, Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ, αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση του μπλοκ αυτού. Ψηφίσατε όλοι. Die Abstimmung ist Πέρας ψηφοφορίας. Abgelehnt ε, Απορρίπτεται. Το μπλοκ ε, Γ, σε υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. D. Ο συνάδελφος πίσω ζήτησε το λόγο ε, επί του κανονισμού. Σε ποιο άρθρο αναφέρεστε παρακαλώ. Πρόεδρε, γιατί θα ψηφίσουμε έτσι. Εγώ διαφωνώ στις διάφορες τροπολογίες. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσω υπέρ ή κατά. Υπάρχουν τροπολογίες στα μπλοκ που υπερψηφίζω και άλλες καταψηφίζω. Αυτό είναι παρεμπόδιση και παρακόλληση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και του δικαιώματος ε, άσκησης ε, της ελευθερίας του βουλευτή. Ο κύριος Γιούρεκ. Πρόεδρε, εγώ καταψήφισα την ιδέα του να ψηφίσουμε ομαδικά τις τροπολογίες. Αλλά εφόσον το αποφασίσαμε και αν υπάρχουν ονομαστικές ψηφοφορίες εντός του μπλοκ, τότε θα πρέπει να ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση όλο το μπλοκ αυτό, όλη την ομάδα αυτή των τροπολογιών. Έτσι, με ονομαστική κλίση. Κύριε Γιούρεκ, και γιατί δεν μαρτύρεστε, δεν καταλαβαίνω. Μέχρι τώρα δεν ψηφίσαμε κανένα μπλοκ που να ζητούσε ονομαστική ψηφοφορία. Και ακριβώς αυτό θα σας πρότεινα τώρα, το μπλοκ D, να το ψηφίσουμε συνολικά ονομαστικά. Και αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Abgelehnt. Απορρίπτεται. Μπλοκ ε έχει επίση ονομαστική, άρα ψηφίζουμε ολόκληρο το μπλοκ ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και αν ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μπλοκ F. Ονομαστικά και αυτό αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία.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 καταπίπτουν. Συνολική ψηφοφορία τελική, ονομαστική και αρχίζει τώρα παρακαλώ.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 Θα ήθελα να σας πω ότι και το Block G διεκπαιρεώθηκε και κατέπεσε εφόσον εγκρίθηκε προηγούμενο. Πάμε τώρα στην έκθεση Van Den 307 και 423 ονομαστικά ταυτίζονται αυτές οι δύο Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Εάν ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Διαφωνείτε να ψηφίσουμε πάλι έτσι με μπλοκ τις τροπολογίες. Ο κύριος συνάδελφος. Ευχαριστώ. Θα υπήρχε η δυνατότητα, μια που θα ψηφίσουμε unblock, να κάνουμε όλες τις, ε, τις ψηφοφορίες ηλεκτρονικά. Όχι μόνο εκεί που λέει ονομαστική, να τις κάνουμε όλες ηλεκτρονικά από την αρχή. Βεβαίω, με χαρά, αγαπητέ συνάδελφε. Λοιπόν, το πρώτο μπλοκ. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το δεύτερο μπλοκ. Ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, όχι. Τώρα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το τρίτο μπλοκ, C. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Μπλοκ D. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Μπλοκ ε. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. F ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ε, ε τα μπλοκ G και H τώρα καταπίπτουν και θα ψηφίσουμε το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά. Αρχίζει τώρα παρακαλώ η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση Ερτούκ. Οι τροπολογίες 290 και 308 είναι ταυτόσιμες. Αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. μου. Πέρασε. Απορρίψετε. Το μπλοκ Α. Ο κύριος Στεχόφσκι ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Πρόεδρε, για το άρθρο 182α. Είμαι κατά. Είμαι κατά του τρόπου που διενεργείται την ψηφοφορία. Για λόγους που θα υποβάλω γραπτός στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι παραβιάζονται διάφοροι κανόνες με τον τρόπο που δουλεύουμε. Διάφορα σημεία του εσωτερικού κανονισμού. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό το πρόβλημά μου. Ευχαριστώ, το λαμβάνω υπόψη. Μπλοκ Α, ονομαστικά. Ε, Άρχιτε ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Πέρασε. Μπλοκ Β. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Haben alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Βλοκ C. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Βλοκ D. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Μπλοκ ε, ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Άρα τα μπλοκ F και G εμ, καταπίπτουν και ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία. Τελική είναι αυτή. Μάλιστα. Ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι.